δημοσιευτούν μαζί με τις, τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίας, αυτές οι 12 πράξεις. Έρχομαι λοιπόν στη σημερινή ημερήσια διάταξη βάσει του άρθρου 149 της ημερήσιας διάταξης ενέκριναν ε, οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων το σχέδιο οριστικής ε, ημερήσιας διάταξης. Θέλετε να λάβετε το λόγο για διαδικαστικό θέμα τώρα. κανόνα 32 για τη σύνθεση των πολιτικών ομάδων, Πρόεδρε. Δεν ε, μα ενημερώσατε για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση στη σύνθεση των πολιτικών ομάδων. Στην τελευταία σύνοδο σα είχα ρωτήσει αν η κυρία Τζάνι Άτκινσον ε, έχει ε, εκδιωχθεί από την ομάδα του EFDD. Γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο το κόμμα UKIP λέει ότι εκδιώχθηκε από το κόμμα. Ο πρόεδρος του, ε, της ομάδας του EFTD ε, είπε στην τελευταία μας συνεδρία ότι εκδιώθηκε πράγματι. Όμως ο ε, κανόνας 32 δεν προβλέπει αναστολή. Ε, συγγνώμη, είχε, μας είχε δηλωθεί ότι είχε αναστολή ταλή ιδιότητα του μέλους της. Δεν προβλέπεται αναστολή από τον κανόνα 32. Ε, το, το μέλος αυτό κατηγορείται για απάτη. Εδώ ε, ε λαθρέα παραμένει στην ε, ομάδα του EFTD παρόλο που στο ΕΒ δηλώνουν ότι εκδιώχθηκε. Μπορεί να γίνει κάτι για αυτήν την υποκρισία κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κόρμπετ. Μέχρι στιγμής δεν βρήκα κανένα άρθρο του κανονισμού που μου δίνει τη δυνατότητα να δράσω κατά της υποκρισίας. Θα ελέγξουμε όμως αν ο πρόεδρος έχει πράγματι κάποια δυνατότητα να δράσει κατά της κοινοβουλευτικής υποκρισίας. Κατά τα άλλα, καμία πολιτική ομάδα δεν μου έχει κάνει μια σχετική ανακοίνωση για τη συνάδελφο που αναφέρεται ούτε σε σχέση με μια αναστολή της συμμετοχής στην ομάδα είτε σε σχέση με μια ενδεχόμενη εκδίωξή της. Ούτε εγώ ούτε οι υπηρεσίε μου γνωρίζουν κάτι σχετικό. Κύριε Άντριου, θέλετε το λόγο. Άγνιου μάλλον. Yes, uh, I would like Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω τα όσο υπόθηκαν. Η κυρία Άρκινσον εκδιώθηκε υποτίθεται και μάλιστα έγινε και μία έθεση, μία προσφυγή, η οποία δεν έχει ακόμα εκδικαστεί. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση μέχρι να έχουμε μία οριστική απόφαση ανήκει στην ομάδα μας, συμμετέχει στην ομάδα μας. Okay, Ευχαριστώ κύριε Άγνιου, το καταγράφουμε και φυσικά και ο κύριος Κόρμπετ το έχει ακούσει για την Δευτέρα, για τη σημερινή συνεδρίαση. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις αλλαγής της σημερινής διάταξης, όχι. Οι πράσινοι για την τρίτη τώρα έχουν ζητήσει να υπάρξει μια δήλωση της Κομισιόν σε σχέση με την παρακολούθηση πολιτικών, δημοσιογράφων, πολιτών κτλ. της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ε, Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας NSA των Ηνωμένων Πολιτειών ζητά να τεθεί μετά από την ε, έκθεση Μακοβέη στην ημερησία ένταξη της Τρίτης χωρίς ψήφισμα. Εάν γίνει δεκτή αυτή η αίτηση όμως, πρέπει να σας πενθυμίσω ότι η προφορική ερώτηση για τα λεγόμενα FEE e σύνορα θα πρέπει να αναβληθεί για την πρώτη συνεδρία σε Ολομέλειας του Μαΐου. Η κυρία Χάρμ για να υποστηρίξει την πρόταση των Πρασίνων. Παρακαλώ κυρία Χάρμ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. όταν βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα οξύ σημείο σε σχέση με την υπόθεση της NSA, ε, είχε πει η κυρία Μέρκελ ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια μορφή κατασκοπίας. Αλλά είναι φανερό ότι υπήρξε κατασκοπία συμμάχων και φίλων από την NSA μέσω και της Γερμανικής Υπηρεσίας Συλλογής Πληροφοριών, ενδεχομένω και μέσω άλλων υπηρεσιών συλλογής πληροφοριών που έχουν γίνει υποχείρια της NSA. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε πώς θα, θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα τέτοιο καυτό θέμα ε, κατασκοπίας εναντίον πολιτικών, εναντίον επιχειρήσεων, εναντίον πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι δεν θέλουμε να περιμένουμε και να αφήσουμε να περάσει αυτό το γεγονός. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η νέα διάσταση που έχει αναλάβει η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφαλείας, η NSA, απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιδράσει και γι' αυτό ζητούμε να τεθεί στην ημερήσια διάταξη. Μετά από την κυρία Ένστ. Η κυρία Ένστ για την αντίθετη θέση αλλά για την υποστήριξη αυτού του θέματος. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτό το σημείο. Η NSA έχει χρησιμοποιήσει ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών για να πάρει πληροφορίες από επιχειρήσεις. Αυτό όμως αποτελεί πραγματική εμπορική κατασκοπία που απαγορεύεται από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης υπήρξε κατασκοπία πολιτικών και απλών πολιτών με εντολή της NSA. και επομένως είναι φανερόν ότι έχει παραβιαστεί το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανονισμοί και οδηγίες που έχουμε εγκρίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο, δεν μπορούμε να το, να το αποδεχτούμε. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και πιστεύω και οι άλλες ομάδες πρέπει να συνενέσουν σε αυτή την ε, αντιμετώπιση. Ευχαριστώ, λέει ο Θέλει κάποιος να λάβει το λόγο κατά της αίτησης της κυρίας Χάμς. Όχι. Οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε για την αίτηση της κυρίας Χάμ και των Βασίλου. Ποιο είναι υπέρ αυτή τη πρόταση. Κατά. Αποχές. Ίσως πρέπει να, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά κυρίε και κύριοι. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι και όλες, αγαπητοί συνάδελφοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 187 υπέρ, 127 κατά, 9 αποχές. Γίνεται δεκτή λοιπόν η αίτηση αυτή της κυρίας Γάμπης και των Πρασίνων. Επίσης στην Τρίτη υπήρξε μια αίτηση της ομάδος της GUE NGL να συμπεριληφθεί μια δήλωση της Κομισιόν για την κατάλληλη προστασία των ε, καταγγελόντων και των δημοσιογράφων σε σχέση με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Για την υποστήριξη, χωρίς ψήφισμα μάλιστα, για την υποστήριξη του θέματος αυτού έχει το λόγο ο κύριος Δεμάση. Κύριε Πρόεδρε, ο Εντουάρτ Περέ, ο Γάλλος αυτός ε, δημοσιογράφος, αυτή τη στιγμή κατηγορείται στο Λουξεμβούργο για την ανάμειξή του στην υπόθεση LuxLeaks. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης, θέλουμε όμως να σεβαστούμε και την ε, προστασία των δημοσιογράφων και την ανεξαρτησία του τύπου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει προστασία των ε, καταγγελόντων και των δημοσιογράφων δεν έχει νόημα σε επίπεδο δικαίου όταν αυτοί οι οποίοι διώκονται δεν είναι οι υπεύθυνοι, αλλά για αυτοί που τα αποκαλύπτουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον κύριο Γιούνκερ, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για το Λουξεμβούργο πάρα πολλά χρόνια, θα πρέπει να έρθει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υποβάλει προτάσει για ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και η αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον αγώνα κατά τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να υποστηρίξει αυτήν την αίτηση, ε, ε, ο κύριος Λάμπερτς. Κύριε Πρόεδρε, ε, χωρίς ε, το, το καμπανά κινδύνου εκ μέρους του δεν θα είχαμε την τροπολογία που είχαμε, δεν θα είχαμε το πακέτο που είχαμε κλπ. Οπότε είναι σημαντικό να ενθαρρύνουμε αυτούς οι οποίοι καταγγέλουν ε, και η Κομισιόν στο δεύτερο ε, φορολογικό της πακέτο θα πρέπει να περιλάβει διατάξεις για να προστατευθούν αυτοί οι καταγγέλλοντες. Δεδομένων των τελευταίων γεγονότων, πιο πρόσφατων γεγονότων, είναι απαραίτητο. Θέλει κάποιος να, λάβει το λόγο κατά αυτής της πρότασης. Όχι. Μπορούμε να ψηφίσουμε λοιπόν. Ποιος είναι υπέρ της πρότασης του κυρίου Ντιμάτση και Γκουε, παρακαλώ. Κατά αποχές γίνεται δεκτή αυτή η αίτηση. Δεν έχω άλλε αιτήσει για την Τρίτη. Περνάμε στην Τετάρτη. Η Σοσιαλιστική και Δημοκρατική Ομάδα ζήτησε μια δήλωση, να συμπεριφθεί μια δήλωση τη Αντιπροέδρου τη Επιτροπή και υπά τη εκπροσώπου για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση για, σε σχέση με την κατάσταση του Μπουρούντι να προσθεθεί ως πρώτο σημείο στην ημερήσια διάδοξη Τετάρτη χωρί ψήφισμα. Η κυρία Κιέγγι έχει το, το λόγο πρώτα για να παρουσιάσει αυτή την αίτηση. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματο ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θέλουμε μία δήλωση τη ύπατη εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξωτερικέ υποθέσεις, δηλαδή από την κυρία Μογκερίνη, προκειμένου να συζητήσουμε εδώ πέρα στην Ολομέλεια τόσα συμβαίνουν στο Μπουρούντι, ιδίω μετά την υποψηφιότητα για τρίτη εντολή του Πρόεδρου Κουμουσίζα. Πρέπει να σα υπενθυμίσω ότι τι τελευταίε αυτέ ημέρε, μετά την υποψηφιότητα αυτή, η οποία τίθεται κατά των συμφώνων τη ΑΟΣΑ για την ειρήνη, πολύ φοβόμαστε ότι η ειρήνη στην όλη περιοχή ενδεχομένω να τεθεί εν κινδύνο και κατά αυτόν τον τρόπο να αποσταθεροποιηθεί όλη η περιοχή των μεγάλων λιμνών. Θέλουμε λοιπόν μια δήλωση χωρί ψήφισμα προκειμένου να δούμε ακριβώ πώ έχει κατάσταση στην περιοχή. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιο να λάβει το λόγο υπέρ αυτή τη αίτηση. Κύριε Λάμπερτς. Υποστηρίζουμε αυτό το αίτημα. Πολύ δε περισσότερο που είναι πολύ επίγον. Αν αναβληθεί ε, θα είμαστε πολύ πιο κοντά στις εκλογές. Οπότε την υποστηρίζουμε. Κάποιος θέλει να λάβει το λόγο κατά αυτής της αίτησης. Όχι. Ψηφίζουμε τότε. Ψηφίζουμε την αίτηση της κυρίας Κίνγκη. Ε, ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Γίνεται δεκτή η αίτηση. Επίσης την Τετάρτη η ομάδα του ΕΛΚ έχει ζητήσει η ζήτηση για τον για θανάτωση φοιτητών στην Κένια να παρουσιαστεί με ένα διαφορετικό τίτλο ε, «Δίωξη χριστιανών σε όλο τον κόσμο σε σχέση με τον φόνο φοιτητών στην Κένια από την τρομοκρατική ομάδα Al-Shabaab». Ο κύριος Φέμπερ για να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλουμε να αλλάξουμε τον τίτλο όπως αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο για να προσθεθεί η έννοια των χριστιανών και της δίωξης των χριστιανών με εκπεφρασμένο τρόπο για δύο λόγους. Καταρχήν είναι αυτό το γεγονός στην Κένια, γιατί δεν ήταν μονάχα χριστιανοί οι οποίοι εθίγησαν από την βία αυτή αλλά και άλλοι, αλλά η, η βία αυτή υπάρχει μονάχα γιατί υπάρχει το μίσος κατά των χριστιανών που υποδαβλίζεται. Επομένως η πηγή αυτού του γεγονότος είναι ο, το μίσος κατά των ε, χριστιανών. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς θέλαμε να υπάρξει μια αίτηση συζήτηση όχι μονάχα για την Κένια αλλά για τη συνολική κρίση κατά δίωξη κατά χριστιανών. Η Κένια ήταν μονάχα ένα παράδειγμα αυτής της δίωξης. Έχουμε 300 εκατομμύρια χριστιανούς στον κόσμο το από συνθήκες καταδίωξης. 150.000 χριστιανοί χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο. Από την δεκαετία του 1990 από 20% του πληθυσμού οι χριστιανικές μειονότητες έχουν μειωθεί στο 4%. Υπάρχει παγκόσμια πίεση κατά των χριστιανών. Αυτό είναι η μεγαλύτερη λοιπόν, χριστιανή η μεγαλύτερη καταδιωκόμενη θρησκευτική ομάδα, ομάδα στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συζητήσει και ενωμένο να εγκρίνει το ψήφισμα το οποίο ήδη έχει υποβληθεί για το θέμα αυτό της καταδίωξης των χριστιανών σε όλο τον κόσμο και εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι συζητούμε για τα θέματα της δίωξης των χριστιανών, αλλά δεν περιλαμβάνεται αυτό στον τίτλο της ε, συζήτησης. Γι' αυτό ζητώ να τροποποιηθεί ο τίτλος και να λέγεται «Κατά δίωξη των χριστιανών σε όλο τον κόσμο». Με παράδειγμα αυτό της ε, Κένιας. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι ότι επιτέλους μετά από τόσες προσπάθειες της ομάδας μου να υπάρξει μια ευρεία και πλήρη συζήτηση η οποία να ακολουθηθεί από μια ονομαστική ψηφοφορία. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Ποιος θέλει να υποστηρίξει αυτήν την αίτηση. Ποιος θέλει να λάβει το λόγο υπέρ αυτής της έτσι; Παρακαλώ. Ε, κυρίες και κύριοι, στηρίζω αυτή την ιδέα. Θα πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Πρόκειται για διώξεις κατά χριστιανών. Διώξεις εδώ σε αυτή τη μεριά του κόσμου. Σε άλλες μεριές του κόσμου διώκονται άλλες θρησκείες, αλλά δεν θα πρέπει να αυτολογοκρινόμαστε. Στηρίζω το αίτημα. Er ο κύριο Γκερέρο θέλει να λάβει το λόγο κατά αυτής της αίτησης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να διακρίνω το θέμα τη δίωξη των χριστιανών ε, από το συγκεκριμένο θέμα της ε, τρομοκρατικής επίθεσης στην Κένια. Πρόκειται για μια αδιαφεσβήτη πραγματικότητα ότι οι χριστιανοί σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερως ε, στην Μέση Ανατολή, υπόκεινται σε συνεχείς διώξεις δραματικές για δύο συγκεκριμένους λόγους. Πρώτον, εξαιτία του αριθμού των θυμάτων και δεύτερον, επειδή πρόκειται για προγραμματισμένη δράση, ε, σχεδιασμένη δράση με στόχο να εκριζωθούν οι χριστιανοί από την περιοχή αυτή και να εξαφανιστούν οι κοινότητές τους. Οπότε συμφωνώ ότι πρόκειται για ένα δραματικό ζήτημα, ένα τραγικό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται να το δούμε με νυφαλιότητα. Η ομάδα μου συμφωνεί το συντομότερο να συμμεριληθεί στην μερίσια διάταξη ε, της ε, Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το συντομότερο λέω, στην επόμενη σύνοδό μας να συμπεριλάβουμε μια συζήτηση για τη δίωξη των χριστιανών για τις διώξεις των χριστιανών. Ε, όμως, για το θέμα της επίθεσης στην Κένια, όπως γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, στην διάσκεψη των Προέδρων ε, ε αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε τη λέξη Ισλαμικό Ισλαμική ε, που βρισκόταν αρχικά στον τίτλο προκειμένου να μην δημιουργήσουμε την αίσθηση ε, θρησκευτική σύραξης. Ε, μάλιστα το ΕΛΚ ζήτησε αργότερα να μπει το ζήτημα των διώξεων των χριστιανών. Δεν πιστεύω ότι είναι σωστό γιατί κάποιοι από τους θανόντες άλλωστε δεν ήταν χριστιανοί. Οπότε προτείνουμε ως ομάδα μια συζήτηση για τις διώξεις των χριστιανών στον κόσμο σε μια επόμενη σύνοδο της Ολομέλειας και να μην αλλάξουμε τον τίτλο της συγκεκριμένης τρομοκρατικής επίθεσης στην Κένια. Εντάξει, <clears throat> ευχαριστώ λέει Έχουμε λοιπόν την αίτηση του κυρίου Βέμπερ και ακούσαμε τις δύο θέσεις υπέρ και κατά. Έχει ζητηθεί ονομαστική κλίση για την αίτηση αυτή. Άρχεται λοιπόν η ψηφοφορία ηλεκτρονικά και ονομαστικά. Άρχεται. Haben alle und Kollegen abgestimmt. Έχετε ψηφίσει όλες και όλοι. Επαναλαμβάνω, ψηφίσατε όλες και όλοι, πέρα στις ψηφοφορίες. γίνεται δεκτή. Ψήφισαν 192 υπέρ, 134 κατά, 13 αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν η αίτηση αυτή. Δεν έχω περαιτέρω αιτήσει τροποποίηση τη ημερήσια διάταξη. <clears throat> Επομένω, έχει οριστικοποιηθεί η ημερήσια διάταξη. Το επόμενο σημείο είναι η